Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την ε, συνεργασία σας. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη Ολομέλεια του Μαΐου. Και τώρα πάμε στην επόμενη συζήτηση. Προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την απαγόρευση της εξόρυξης ε, ε τεχνολογιών, εξόψη συγγνώμη μετάλλων ε, με τεχνολογίες που βασίζονται στη χρήση κυανιούχων ενώσεων. Ο κύριος ε, Ζάνος Αντέρ. Τρία λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Τα τελευταία χρόνια έχουν ε, ληφθεί πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος και ήθελα να αναφερθώ στις αποφάσεις που αναφέρονται ή στη βιοπικιλότητα ή ε, την ε, οδηγία, για, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, για την προστασία των υδάτων μας και για να αποφύγουμε τη ρήπανση των υδάτων. Αυτός δεν είναι ο στόχος που επιζητούμε, ναι αλλά ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Και αυτό αναφέρεται εις ε, την εξορρυκτική πρακτική η οποία θέτει σε κίνδυνο τη βιοπικιλότητά μας και υπάρχει μια τέτοια πρακτική η οποία ε, θέτει σε κίνδυνο την ε, κατάσταση. Θα έπρεπε λοιπόν να απαγορεύσουμε αυτή την τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι πριν από 10 χρόνια η καταστροφή από Κιανίδιο εις το ποτάμι Τίσα ε, ε, προκάλεσε τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της κεντρικής Ευρώπης και το θέμα παραμένει επίγον διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο τρεις χώρες χρησιμοποιούν τεχνολογία που βασίζεται και τρεις άλλες ε, χώρες έχουν ήδη ε, απαγορεύσει αυτή ε, την τεχνολογία θέτοντας ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Κατόπιν αυτού αυξάνεται όμως η τιμή του χρυσού και μπορεί να ανοίξουν και νέα χρυσορυχεία οπότε υπάρχει πάρα πολύ οξύ κίνδυνος για το περιβάλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν εννοούμε αυτό που λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα των υδάτων μας, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε αυτές τις ουσίες δίπλα στα ποτάμια μας και ε, να ε, συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πεπαλαιωμένες τεχνικές. Πρέπει ε, να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, να μην σκοτώνουμε τη ζωή που υπάρχει μέσα στο νερό από ψάρια, από στρακοειδή και θα έπρεπε να μην περιμένουμε να έρθει μία νέα καταστροφή για να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα του θέματος. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και να υποφεληθώ για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, οι οποίοι συνεργάστηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω του ηφαιστείου και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ε, ε, στήριξη στην συμβιβαστική πρόταση που στηρίζεται και από το ΕΛ και από τους σοσιαλιστές και από τους φιλελεύθερους και από τους αριστερούς καιρούς οπότε σας παρακαλώ να συνεχίσετε να μας στηρίζετε μέχρι να υιοθετηθεί η συμφωνία. Ευχαριστώ στην η κυρία Μάλστρο με ονόματι της Επιτροπής. Αγαπητοί βουλευτές, ο κύριος Πίμπαλκ, ο συνάδελφός μου ε, σας ζητάει συγγνώμη, δεν θα μπορέσει να παραστεί ε, και μου ανέθεσε το καθήκον να εκφράσω την άποψη της Κομισιόν. Ε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να χρησιμοποιήσω τη θέση της ε, Κομισιόν για τη χρήση του, κιαν, του κιανίου στην εξορρυκτική βιομηχανία. Όπως γνωρίζετε, ε, είχαμε μία πολύ, ετοιμάσαμε μία πολύ σοβαρή μελέτη ε, για το ατύχημα που έγινε στη Ρουμανία το 2000 ε, όταν απορρίφθηκαν τέτοιες ουσίες σε ποτάμια. Για το 2000 ε, υιοθετήσαμε μία οδηγία για την διαχείριση των αποβλήτων από την εξορρυκτική βιομηχανία. Ε, το όριο για τη μετάθεση στην εσωτερική νομοθεσία ε, ήταν δύο χρόνια, πριν δύο χρόνια. Η οδηγία έχει διάφορες προϋποθέσεις για να αυξηθεί η ασφάλεια για τη διαχείριση των αποβλήτων, συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την κατασκευή των τόπων διάθεσης που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις καλύτερες τεχνικές. Ε, υπάρχει μια πολιτική ε, για την πρόληψη εκεί όπου αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται τις τοξικές ε, ουσίες. Και θα πρέπει να έχουν και σχέδια κατεπήγοντος και οι αρμόδιες αρχές αλλά και οι εγκαταστάσεις αυτές. Επίσης, ε, προϋποθέσεις ενημέρωσης, εάν υπάρχουν και επιπτώσεις διασυνοριακές. Αυτή η νομοθεσία, επίσης, έχει και προϋποθέσεις για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και τι γίνεται μετά το κλείσιμο. Και πριν αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι εγκαταστάσεις υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν ε, ανώτατα όρια ε, των οριακών τιμών για τις συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών πριν αποθηκεύσουμε σε τεχνητές λίμνες αυτές τις ουσίες για να τις διασπάσουμε με την οξύδωση κτλ. Ε, πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένο ε, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένους μηχανισμούς. Από ό,τι γνωρίζουμε, δυστυχώς όμως, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση κιανίου στα χρυσορυχεία. Εσύ, σε περισσότερες περιπτώσεις χρειαζόμαστε μια μέθοδο διαχωρισμού του χρυσού από τα άλλα μέταλλα. Ε, αν δεν χρησιμοποιήσουμε κιάνιο, ε, θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε να εξορίσουμε χρυσό και θα αναγκαστούμε να τον εισάγουμε από το εξωτερικό, ε, με όλες τις ε, επιβαρύνσεις. Ε, Βεβαίω γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξελίξει στην τεχνολογία και αν υπάρξουν εναλλακτικέ τεχνικέ τα επόμενα χρόνια μπορεί να ξανανοίξει η συζήτηση. Στο μεταξύ όμω, μια καλή εφαρμογή αυτή τη οδηγία είναι εκ των ονουκάνευ για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων και να μειώσουμε τον κίνδυνο που συνδέεται με τη διαχείριση. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι πάνω απ' όλα τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για να αποφασίσουν να ανοίξουν χρυσορυχία στο εδαφό του. Ο ρόλο τη Κομισιόν είναι εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τη οδηγία και, την εφαρμογή, και η σωστή εφαρμογή είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν. Με βάση την οδηγία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν στην Κομισιόν πληροφορίες για την εφαρμογή ε, το αργότερο το 2012. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την αναλύσουμε, τις αναλύσουμε τις πληροφορίες και να ε, καταρτήσουμε μία έκθεση. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης. Αν αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι αποτελεσματική, δεν αποκλείεται να αλλάξουμε μέθοδο. Ε, θέλουμε να έχουμε υψηλό επίπεδο ανακύκλωση των αποπλήτων και αποτελεσματικότητα στην εξοριξτική βιομηχανία. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η εξόριξη ε, χρυσού είναι κακή ε, για το περιβάλλον. Καταλαβαίνουμε ότι για να εξορίξουμε μόνο ένα γραμμάριο χρυσού ε, πρέπει να εξορίξουμε πολύ περισσότερα μεταλλεύματα. Ξέρουμε πολύ καλά επίσης τι, απόβλητα ε, απορρίπτουμε στο περιβάλλον. Ε, η αποτελεσματικότητα λοιπόν αυτής της βιομηχανίας είναι προτεραιότητα της ε, Επιτροπής μας. Ε, τώρα, οι πολιτικές ομάδες, ο κύριος Σίμπερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι διότι ε, εδώ θα προτιμούσα να είχα εδώ τον κύριο Ποτότσνικ διότι αυτό είναι που θα πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα διότι ξέρω ότι η Ευρώπη έχει μία παραγωγή χρυσού κάτω από το 1% και υπάρχει εξόριξη ε, του χρυσού στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, σε διάφορες χώρες ε, χρησιμοποιώντας όχι πολύ σύγχρονη τεχνολογία. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αφενός υπάρχουν κατάλληλες αντιλήψεις για την αποθήκευση των εξορυκτικών υλικών και επίσης ότι οι αρχές που έπρεπε να επιτηρούν δεν παρακολουθούσαν επαρκώς τα μεταλλεία. Δηλαδή υπήρχε συσσόρευση πορών λαθών και όπως είπε και η Επίστροπος ε, διδαχθήκαμε από το ατύχημα αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε και σε άλλα ε, συμπεράσματα. Εφόσον λοιπόν οι τεχνολογίες τις οποίες έχουν δεν δίνουν το ε, αποτέλεσμα το οποίο αναμένουμε πρέπει να δούμε τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε καταρχήν την περαιτέρω εξόριξη χρυσού αλλά και την ασφαλή καλή εξόριξή του. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζουμε τις ε, ασφαλείς προδιαγραφές και ε, να σεβόμαστε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την βιοπικιλιότητα. Οπότε γι' αυτό θα θέλω να παρακαλέσω την Επίτροπο να συνεχίσει να υπαγνυπνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα της εξορίξεως χρυσού. Ευχαριστώ κύριε Σίμπερ και το λόγο έχει κύριος Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Εμείς ως ε, χριστιανοδημοκράτες υποστηρίζουμε, στους δημοκράτες μάλλον, υποστηρίζουμε την απαγόρευση της χριστιανίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θέλω να υπογραμμίσω, κυρία Επίτροπε, και να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι δεν είναι να παίρνετε αναδρομική δράση. Δυστυχώς στην Ευρώπη η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε δει αυτό στην Επιτροπή Αναφορών. Υπάρχει ρήπανση, προσπαθείτε να δράσετε εκ των υστέρων. Δεν είναι πρόληψη αυτό. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να ξεκινήσουμε με την πρόληψη. Ο κύριος Άκερ και ο κύριος Ζέμπερ ανέφεραν την ε, καταστροφή του Μααμάρε. Όταν λοιπόν ζητάμε την απαγόρευση της χρήσης κυανούχων ουσιών για την εξόρυξη μετάλλων, βασιζόμαστε σε μια θλιβερή προηγούμενη εμπειρία. Στη Ρόζε Μοντάνα έχουμε πολύ μεγάλα χρυσορυχία σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και εκεί αντιμετωπίζεται μια σωρία προβλημάτων στο σχέδιο αυτό. Δεν υπάρχει παραμικρή εγγύηση ότι η τεχνολογία ανοιχτή εξόρυξης, ανοιχτών ορυχείων δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον γιατί διαβρώνουν οι δηλητηριώδεις και οι ανήρχες ουσίες στον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον και δεν υπάρχει λοιπόν καμία εγγύηση ότι όταν θα τελειώσει η εξορυκτική δραστηριότητα θα μπορέσει να ε, αποκατασταθεί το τοπίο στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και, σοσιαλιστές και Δημοκράτες μα με την ΚΟΕ και τους Πράσινους και την Ελεύθερη Συμμαχία ζητούμε από την Κομισιόν να αναπτύξει νομοθετήματα μέχρι το 2011 ώστε να υπάρξει οριστική χρήση οριστική απαγόρευση της χρήσης ανιούχων ουσιών στην εξόρυξη. Γιατί η ρήπανση δεν μπορεί να σταματήσει στα σύνορα μερικών χωρών. Δεν αρκεί μερικέ μοναχα χώρες να την απαγορεύσουν αυτή την τεχνολογία δεν υπάρχει συνολική λύση. Ο κύριο Τρεμόπουλο για ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητούμε γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο υλικό το κυάνιο. δεν αποδεχόμαστε αυτό που ακούσαμε από την εκπρόσωπο της επιτροπής ότι δεν υπάρχουν ε, μη επικίνδυνες τεχνικές. θεωρούμε ότι στην ελλάδα από τη στιγμή που υπάρχουν τρία επενδυτικά σχέδια μεταλλουργίας χρυσού με κυάνιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την απαγόρευση αυτής της τεχνικής στον εύρο στη ροδόπη στη χαλκιδική υπάρχει αντίδραση στεναρή των τοπικών κοινωνιών και υπάρχουν και αποφάσεις από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο το συμβούλιο της επικρατείας της χώρας. η απειλούμενη εμπλοκή του διεθνούς νομισματικού ταμείου λόγω της κρίσης στη χώρα μου δημιουργεί φόβους και για πιθανές πιέσεις και χαλάρωση της νομοθεσίας που προστατεύει το περιβάλλον αλλά και των ελέγχων. υπάρχουν πρακτικές και εμπειρίες από άλλες χώρες με τραγικά αποτελέσματα. στην ελλάδα οι κίνδυνοι προέρχονται και από ε, εκμετάλλευση χρυσού στη βουλγαρία που είναι στην λεκάνη απορροής του εύρου. επίσης υπάρχει ζήτημα με τα παράλια της τουρκίας και απειλές για το αιγαίο. υπάρχουν τέτοια σχέδια και σε άλλες χώρες. η ουγγαρία όμως όπως ήδη γνωρίζουμε μόλις το δεκέμβριο αποφάσισε την απαγόρευση όλων των μεταλλουργικών διεργασιών που βασίζονται στο κιάνιο. θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρη απαγόρευση και ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός δικτύου ε, ασφαλείας για χώρες ευάλωτες οικονομικά όπως η ελλάδα. ζητούμε η αδύναμη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης να γίνει πιο αποφασιστική και να μην υπάρξουν πια διαφορετικά επίπεδα στους επιτρεπόμενους ρήπου ανά κράτος μέλος. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόπουλε. Ο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς θέλω να πω ότι το θέμα το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και δεν χωρούν κολυσιεργίες. η επιτροπή και η στάση που έχει κρατήσει είναι χαλαρή η οδηγία είναι διάτρητη δεν εξασφαλίζει τους κινδύνους δεν αποτρέπει τους κινδύνους στους οποίους αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι. είναι γνωστή η σημασία και οι επιπτώσεις που έχει η χρήση του κυανίου στην εξόρυξη μετάλλων έχουμε το παράδειγμα της ε, ρουμανίας. ο συνάδελφος που προηγήθηκε αναφέρθηκε σε εξορυκτικά προγράμματα που εκπονούνται αυτή την περίοδο στην ελλάδα σε σχετική ερώτησή μου στην επιτροπή σε σχέση με τη δημιουργία μεταλλείου χρυσού με τη χρήση κυανίου στη βουλγαρία η απάντηση της κομισιόν ενίσχυσε τους φόβους μου και την ανάγκη αυτή η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή και η εφαρμογή της πιο αποφασιστική. είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες προφανώς θα αντιδράσουν αλλά θα πρέπει να ενεργήσουμε. ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μα μαζί με όλου όσου ζητούν την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου ε, για την εξόριξη πολυτήμων μετάλλων και θα πρέπει όλες οι χώρες όπως πρόσφατα έκανε η ουγγαρία να δεσμευτούν σε αυτή την απαγόρευση. σας ευχαριστώ. λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προασπίζονται την υγεία, τη φύση και ε, την βιοπικιλότητα προς τα έξω. Είναι λοιπόν περίεργο ότι ε, στην περίπτωση αυτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ευρωπαϊκές διατάξεις διότι είναι γνωστό ότι τα κιανίδια είναι από τις πιο επικίνδυνες τοξικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν και να βλάψουν την, ε, ε, το δέρμα και ε, να μπορέσουν να οδηγήσουν στο θάνατο χρυσορίχους εντός λεπτών και τα μέτρα προστασίας δεν έχουν γίνει σεβαστά. Μας εκπλήσει λοιπόν η φύση και και βλέπουμε πολλές ε, περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι υπήρξαν ατυχήματα που οδήγησαν και σε απώλειες ζώων ακόμη και τα τελευταία εις το Κολοράντο ή στην Νότιο Καρολίνα ή στην Νότιο Αφρική ή στην Εβάδα ή στο, στη Μοντάνα, στην Αμερική ή στην Νότιο Ντακότα ή στις Φιλιππίνες, Ρουμανία και στη Βαπούα Νέα Γουινέα και στις περιπτώσεις αυτές και το περιβάλλον ε, και, το, ε, ε, και οι άνθρωποι πλήρωσαν ένα υψηλό τίμημα για τις ρηψοκίνδυνες αυτές πρακτικές των χρυσορίχων και θα πρέπει να φροντίσετε να προστατεύσετε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών μας και να μην προσπίζετε τα συμφέροντα των χρυσορίχων. Ο κύριος Στανασέσκου για δύο λεπτά τώρα. Ευχαριστώ. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το κιάνιο και η απαγόρευση του κιανίου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος στη Ρουμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι το 2006 έγιναν 25 μεγάλα ατυχήματα, κάτι που αποδεικνύει ότι το ωκεάνιο είναι απειλή για το περιβάλλον που κρατάει εδώ και δεκαετίες. Αυτά τα ατυχήματα έθεσαν ε, τεράστια ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις πρακτικές και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει. Παρότι οι εταιρείε έχουν τις καλύτερες προθέσει βεβαίω. Το ωκεάνιο δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ε, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση αν συνδυάσουμε την κακή διαχείριση με την κακή μέθοδο έχουμε εκρηκτικές καταστάσεις ε, από τη χρήση του κιανίου. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, αλλά δεν τις προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η προώθηση αυτή θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί, γιατί υπάρχουν πραγματικά τεχνολογίες που είναι πολύ πιο σίγουρες. Το, το Νοέμβριο του 2005 οι Ευρωβουλευτές και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για μια οδηγία σε ό,τι αφορά τα απόβλητα από την εξορρυκτική βιομηχανία. Αλλά δυστυχώ αυτό το εργαλείο εξαιτία του λόμπινγκ της βιομηχανίας κατέστη αναποτελεσματική και σε ό,τι αφορά ε, την απροθυμία των χωρών της ε, Κεντρική Ευρώπη, που δεν θέλησαν να ανακυκλώσουν ε, τα παλιά εγκαταλελειμμένα χρυσορυχεία. Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εκπομπή κιανίου στον αέρα. Στη Ρώσα Μοντάνια, στην ε, Ρουμανία, αν ανοίξει αυτή η βιομηχανία, κάθε μέρα θα εκπέμποτε 134,2 κιλά κιανίου στον αέρα. Σε 16 τόσο λειτουργεί ένα χρυσό περίπου θα έχουμε 800.000 ε, κιλά κιανίου στον αέρα. Ποια είναι η ποιότητα του αέρα όταν έχουμε τέτοιες εκπομπές. Έχουμε το δικαίωμα, το και το καθήκον να, για, απέναντι στις επόμενες γενιές να απαγορεύσουμε τη χρήση του κιανίου. Τώρα πάμε στους επόμενους ομιλητές, η κυρία Ρόιτοβα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. μιλάμε για πολύ μεγάλες ε, καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει ιδίω σε χώρες όπως η Ρουμανία. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στην κατάθεση ενός ψηφίσματος το οποίο ζητά μια απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξορρυκτικές δραστηριότητες. Όχι μονάχα είναι επικίνδυνη η χρήση αυτών των ουσιών, αλλά επηρεάζει σημαντικά αρνητικά την φύση. Ένας τόνος κυανούχων ε, ενώσεων μπορεί να, που χρειάζεται για την εξόρυξη ενός γραμμαρίου χρυσού μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια επιβάρυνση της φύσης και των ε, πετρωμάτων στην περιοχή. Λοιπόν, γι' αυτό ζητούμε να υπάρξει υποστήριξη από όλους στην ε, ψηφοφορία για την απαγόρευση αυτής της πλήρους απαγόρευσης των κυριανιούχων ενώσεων από το 2012 για την εξόριξη και να μην υπάρξει πλέον χρησιμοποίηση κυριανιούχων ουσιών. Και προφανώς η Κομισιόν δεν πρέπει να υποστηρίξει κανένα σχέδιο το οποίο χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, Τσεχία, τη Ρουμανία και ε, και τη Γερμανία. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η, η απαγόρευση λοιπόν και δεν μπορούμε εμείς να θέσουμε στην πλάστηκα το κέρδος των εξορρυκτικών εταιρεών έναντι της υγείας των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αρσένης. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Επίτροπε Μάστρομ. Μετά το Τσερνομπίλ κατανοήσαμε όλοι τον πυρηνικό κίνδυνο το 2000 όμως προκλήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης και ίσως παγκοσμίω από το ατύχημα Βάγια Μάρε στη Ρουμανία που αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι. Διέρευσαν από εξωτερική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ ψηλέ συγκεντρώσει κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στο ποταμό Τίσλα και από εκεί στο Δούναβι πλέοντα εκτό από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, σκοτώνοντα δεκάδε χιλιάδε ψάρια και δηλητηριάζοντα το πόσιμο νερό η μόλυνση τροφική αλυσίδα τη άμεσα πληγή σα περιοχή υπήρξε μακροχρόνια. η ουγγαρία ανέφερε 1.367 τόνου νεκρών ψαριών. πάνω από 100 άτομα κυρίω παιδιά δηλητηριάστηκαν και νοσηλεύτηκαν άμεσα έχοντα καταναλώσει τα μολυσμένα ψάρια. παρ' όλα αυτά η εξόρυξη χρυσού με τη χρήση κυανιούχων διαλυμάτων όχι μόνο συνεχίζεται όχι μόνο δεν απαγορεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά οι σχετικέ επενδύσει επιδοτούνται από τα κράτη μέλη και την ευρωπαϊκή ένωση η εξόριξη συνεχίζεται ή προγραμματίζεται να ξεκινήσει στη σουηδία φινλανδία σλοβακία ρουμανία βουλγαρία και στην ελλάδα ενώ απαγορεύεται μέσω νόμου στην ουγγαρία τη τσεχία και μέσω νομολογία στη γερμανία. αγαπητοί συνάδελφοι ο καιρό που ανταλλάσσαμε θέσει απασχόληση, έναντι του τοπικού περιβάλλοντο και τη υγεία των πολιτών ανήκει πλέον στο παρελθόν. ακόμη και η οικονομική βιωσιμότητα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καταρρέει αν εφαρμόζαμε την αρχή της πρόληψης και την αρχή ο πληρώνει. κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι ευπρόσδεκτη εφόσον συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών. όταν όμως χρησιμοποιούμε κιάνιο θέτουμε σε επανόρθωτο κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία των πολιτών. επίτροπε Μάλστρομ είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι έχουμε επαρκή και ισχυρή νομοθεσία και ότι ένα νέο Μπάγια Μάρε δεν θα επαναληφθεί αυτή τη φορά στη σουηδία τη φιλανδία τη βουλγαρία την ελλάδα. αγαπητή επίτροπε ζητώ από την επιτροπή να αποδείξει ότι τιμά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε μόλις πριν από δύο μήνες ενώπιον του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ενώνει τη φωνή μου με τι φωνέ των τοπικών κοινωνιών που υφίστανται πρώτε τι συνέπειε και του αγώνε των περιβαλλοντικών κινημάτων και ζητώ την άμεση απαγόρευση τη χρήση κιανίου για την εξόρυξη χρυσού εντό τη ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ πολύ. Euh, ευχαριστώ κύριε Ασένη. Ο κύριος Κυλακάκης, δύο λεπτά. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, ο χρυσός είναι εκεί δεν πρόκειται να δραπετεύσει. το πότε με ποια τεχνική και ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα αποφασίσουμε να τον εξορίξουμε είναι αυτό που καλούμεθα να συζητήσουμε. αν προχωρήσει μια επένδυση με χρήση κιανίου, οι επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες διότι ο χρυσός φεύγει και τα τέλματα με κυανιούχες επικίνδυνες τοξικές ουσίες κατομολογίαν της ίδιας παραμένουν σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή της εξόρυξης. η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τα κράτη μέλη γιατί υπάρχουν και τα κατάντη κράτη μέλη που βρίσκονται ε, γιατί οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ποταμούς. η υφιστάμενη οδηγία έχει ένα μειονέκτημα η χρηματική εγγύηση που προβλέπεται δεν καλύπτει το σύνολο των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος ιδίως μετά το κλείσιμο των σχετικών εγκαταστάσεων κατά συνέπεια η βασική αρχή ορυπαίνων πληρώνει παραβιάζεται ιδίως με δεδομένο ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική είναι κατά βάση εξωευρωπαϊκές και όταν τελειώνει η εξόρυξη μας κουνούν το μαντίλι και αποχωρούν. θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει μια σοβαρή επανεξέταση των εναλλακτικών μεθόδων εξόρυξης και να αποκατασταθεί η βασική αρχή ορυπαίνων πληρώνει με πλήρη και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη της περίπτωσης ατυχήματος από τώρα και για όσο καιρό παραμένουν αυτές οι επικίνδυνες ουσίες παγιδευμένες στη γη. για όσο καιρό δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση αυτής της τεχνολογίας η οποία θα δώσει ενδεχομένως και κίνητρα για να ερευνηθούν σοβαρά από την πλευρά των εταιριών οι εναλλακτικέ λιγότερο υπογόνες τεχνικές διότι αν έχεις μια φτηνή μέθοδο που δεν πληρώνεις τη ρήπανσή της δεν έχεις λόγο να ερευνάς τις εναλλακτικές δυνατότητες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Σκυλακάκη. Ο κύριος Ρέσνα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αποφάσισα να μιλήσω για το θέμα αυτό σε σχέση με το ψήφισμα ε, κατόπιν ε, των γεγονότων στην Τσεχία ε, όσον αφορά τις μεθόδους με τις οποίες γίνεται η εξόριξη του χρυσού όπου ε, ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων μεταλλεύματος ε, οι οποίες προκαλούν όχι μόνο κυανίδιο αλλά και άλλα οξέα και άλλα τα τα οποία είναι επικίνδυνα και γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχουν μέθοδοι επεξεργασίας μετάλλων ε, χρησιμοποιούνται αυτές οι επικίνδυνες ουξίες οι οποίες ε, ε, θα πρέπει να περιοριστούν σε περαιτέρω εξέλιξη τεχνολογιών αλλά όσον αφορά την εξόριξη χρυσού και τις τεχνολογίες χαίρομαι ότι μετά την απόφαση του 2000 έχει απαγορευτεί η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί και ανίδιο και οι τεχνολογίες αυτές ε, πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς διότι ε, ο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει στις χώρες του τρίτου κόσμου. Κυρία Επίτροπε είσαστε σίγουροι ότι οι νέες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται έχουν λάβει υπόψη ε, τα κινδύνους αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι έθιξαν το θέμα και να σας πω ότι εν πάση περιπτώσει η πρόταση αυτή στηρίζεται ε, ε, εκ μέρους μας για όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια διότι όποιος έχει δει τα αποτελέσματα των περιβαλλοντολογικών ε, καταστραφών όπου μας, δεν μας βοήθησε η τεχνολογία όταν έχουμε δει τις δηλητηριασμένες πηγές όπως στην Ουγγαρία στις πηγές του ποταμού Τίσα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην ξαναυπάρξει κάτι κάτι παρεμφερέσει ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα μου η Σλοβακία έχει πληγεί από αυτές τις καταστροφές οι οποίες έλαβαν χώρα κοντά στα σύνορά μας και ανοίγοντας ορισμένα ορυχεία χρυσού ε, χρησιμοποιήσαμε αυτήν την τεχνολογία ε, που εμπλέκει τη χρήση κιανιδίου. Ε, αυτό δεν είναι ένα διμερές θέμα μεταξύ δύο κρατών κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ελπίζω ότι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα εφαρμοστεί πιο αποφασιστικά από ό,τι μας το παρουσίασε μέχρι τώρα η κυρία Επίτροπος διότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, σε όλη την Ευρώπη τις αξίες μας και να είμαστε συνεπείς στη χρήση των μεθόδων μας. Κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ισορροπημένη θέση που έχει υιοθετήσει και που παρουσίασε στην αρχή α, της συζήτησης. Οι τεχνολογίες με βάση το κιάνιο είναι επικίνδυνες, αλλά και άλλες ε, τεχνολογίες είναι επικίνδυνες, όπως ε, η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Για να εμποδίσουμε τα ατυχήματα υπάρχουν κανόνες και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβαστούμε ε, το, τους κανόνες. Εδώ και 30 χρόνια έχουν συμβεί 25 ατυχήματα. Αποφεύγουμε όμως να μιλάμε για αυτά τα ατυχήματα. Είναι πολύ άριθμα αυτά ε, και κυρίως στις χώρες όπου στο παρελθόν δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το ατύχημα που έγινε το 2000 η νομοθεσία έγινε πιο αυστηρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά για όλες τις τεχνολογίες και στα χρυσορυχεία αλλά και στην παραγωγή φαρμάκων. Το πρόβλημα δεν είναι το κιάνιο ε, αυτό αυτό το πρόβλημα είναι ο χρυσός. Το θέμα δεν είναι να απαγορεύσουμε την τεχνολογία, το θέμα είναι να απαγορεύσουμε δηλαδή όλα τα προγράμματα. Εγώ δεν γνωρίζω άλλες ε, προσπάθειες επεξεργασίας ε, με βάση αυτήν την τεχνολογία πέρα από, αυτό που πέρα από αυτήν στην Ρουμανία. Ε, σας παρακαλώ διαβάσετε το ψήφισμα και Ας προσέξουμε Ας προσέξουμε τι γίνεται με τα χρυσορυχεία. Τα χρυσορυχεία λειτουργούν για 16 χρόνια. Είναι ε, εξορυκτικές βιομηχανίες που ούτως ή άλλως δημιουργούν πολύ λίγες θέσεις εργασίας και μάλιστα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, προσοχή, ε, ας ξαναδιαβάσουμε το κείμενο, να γίνει πιο ισορροπημένο. Θα ήθελα να απορρίψετε αυτό το ψήφισμα γιατί μειώνει την αξιοπιστία μας και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας τις προτάσεις ε, που έχουμε ψηφίσει στο παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρώμος ομιλητής μας είναι η κυρία Νεντέλτσεβα. μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. η χρήση των κυανιούχων ενώσεων δεν πρέπει να αφήνει κανένα αδιάφορο. Έχουμε ήδη αναλάβει κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύσουμε το οικολογικό περιβάλλον με σαφείς και στεναρούς ελέγχους. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε επίσης και την κοινή γνώμη. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με το να πέσουμε με τους φόβους των πολιτών. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν την, τα συμφέροντα συγκεκριμένων εταιριών. Τα, οι ενώσει του κιανίου χρησιμοποιούνται ιδίως στη χημική βιομηχανία και στην επεξεργασία των μετάλλων. Ακόμα και αν υπάρξει απόλυτη απαγόρευση σε σχέση με τη διαδικασία εξόρυξης, αυτό δεν θα σημάνει πλήρη απαγόρευση της χρήσης κιανιούχων ενώσεων σε άλλου βιομηχανικού τομεί. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου στο περιβάλλον τη χρήση ανοιούχων ουσιών και μια αποτίμηση εξ άντε και εξ post σε σχέση με τι κιανουιούχε ενώσει. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απαγόρευση, αλλά δεν υπάρχουν και εναλλακτικέ τεχνολογίες οι οποίες να είναι επαρκώς αποτελεσματικές, ιδίως στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την οδό της λογικής και να μην πέσουμε στις ακραίες λύσεις. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το μεσαίο δρόμο, το δρόμο της Γκαμίλα. Η κυρία Εσάια, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τεχνικές όπως αυτές που οδήγησαν στο ατύχημα της Μπάια Μάρε το 2002. Η Φιλανδία είναι ένας μεγάλος πραγός χρυσού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αρχείο στην Κίτριλα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο, στην Ευρώπη με παραγωγή 5.000 κιλογράμμων χρυσού το έτος. Ένα επιστημονικό γεγονός. Ο χρυσός δεν διαλύεται από κανένα άλλο από καμιά άλλη χημική ουσία εκτός από το υδροκιάνο. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι ανήλικες ενώσεις αλλά σε κλειστά κυκλώματα. Σε διαδικασίες στις οποίες τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται και αφαιρούνται τα υπολείμματα κοινωνιούχων ενώσεων. Γιατί ακόμα και τα απόβλητα στο νερό προτού βγουν από τα φράγματα θα πρέπει να περνάνε μια διαδικασία διήθησης. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες οι οποίες είναι πιο φιλικές προς την, στην, ε, ε στον κόσμο. Δεν χρησιμοποιούνται ακόμα για τον χρυσό. Η μακροβιωτική ε, ο βιωτικός καθαρισμός των ε, λιμάτων από την ε, εξόρυξη χρυσού ήδη χρησιμοποιείται στη Φιλανδία. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον. Εγώ δεν ζητώ την πλήρη απαγόρευση τη χρήση κυανίου ουσιών, αλλά σα ζητώ να χρησιμοποιηθεί η καλύτερη δυνατή υπάρχουσα τεχνολογία και κλειστή διαδικασία κλειστού κυκλώματο για την προστασία του περιβάλλοντο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πρέντα για ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κατά την άποψή μου, το να απαγορεύσουμε το κιάνιο στα χρυσορυχεία και την εξόρυξη του χρυσού δεν δικαιολογείται. Υπάρχουν πολλές πράξεις και πολλές, πολλοί ευρωπαϊκοί νόμοι που αναφέρθηκαν που σκληραίνουν τις προϋποθέσεις χρήσης κιανίου από την εξορυξτική βιομηχανία, βασιζόμενη στα, στην ατυχή εμπειρία, εν του 2000 στην Πάια Μάρε στη Ρουμανία. Νομίζω ότι οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πιο αυστηρή εφαρμογή όλων αυτών των νομοθετικών πράξεων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η τεχνολογία, όπως ε, ακούσαμε ήδη, χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Και τελικά δεν υπήρχαν τόσα πολλά ατυχήματα δεδομένη τη ε, μακροβιότητά τη και είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική για να εξορίξουμε το χρυσό. Ο μεγαλύτερο όγκο ε, χρυσού που εξορίχθηκε στον κόσμο τα τελευταία χρόνια ε, εξορίχθηκε χάρη σε αυτή την τεχνολογία με το κιάνιο. Και πέρα από τους κινδύνους για το περιβάλλον και, και την ανθρώπινη υγεία, στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί χάρη στην πρόοδο τη τεχνολογία. Δεν πρέπει να αντιδρούμε συναισθηματικά. Δεν μπορούμε να, να απαγορεύουμε τα πάντα, ενώ μπορούμε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε του κινδύνου. Η αρχή τη πρόληψη και τη προφύλαξη θα πρέπει να είναι αυτή που πριτανεύει. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που μα λένε οι εμπειρογνώμονε και αν χρησιμοποιούσαμε εναλλακτικέ ε, τεχνικέ, ίσως θα βλάπταμε ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω διάφορους ομιλητές στον κατάλογο. Ο κύριος Τσάμπα Σόγκοριτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy Ευχαριστώ. Η η εξουσιοδότηση για την εξόριξη χρυσού χρησιμοποιώντας κιανίδιο ισχύει σε πολλά κράτη και δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι των πολιτικών συζητήσεων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν οι εμπειρογνώμονες. Αν υπάρχει όντως κίνδυνος ρηπάνσεως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευτούν τα συμφέροντα των πολιτών είναι να αιτιολογήσουμε τεχνολογικά τη χρήση αυτή διότι οι πολίτες δικαιούνται ένα υγιές περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 7 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν λοιπόν ε, κινδυνεύει η υγεία των πολιτών η πολιτική συζήτηση δεν βοηθά και οι αρχές θα πρέπει να αναλάβουν δράση διότι ε, χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ε, χώρες οι ε, μέθοδοι αυτοί με και ανίδιο ενώ αλλού έχουν εγκαταλειφθεί. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να τοποθετηθούν κατά τρόπον ώστε να αποφύγουμε τις δυνητικές βλάβες στην υγεία. Ο κύριος Στακουλέσνα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από ένα υπερβόρειο κράτος στη Φιλανδία και οφείλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Όπως και ο κύριος Εσάια μίλησε ε, και είπε ε, σε μια πολύ καλή παρέμβαση, το κιάνιο χρησιμοποιείται ως διαλύτης στη Φιλανδία σε κλειστά κυκλώματα. Το χρυσορυχείο Κιπτήλα, που είναι πολύ κοντά στην περιοχή που μένω, παράγει πάνω από 5.000 κιλά χρυσού το χρόνο και ποτέ δεν υπήρξαν προβλήματα. Γιατί τα περιβαλλοντικά θέματα τα αντιμετωπίζουμε, ε, έχουμε μοντέρνες διαδικασίες, κλειστά κυκλώματα και η τεχνολογία πραγματικά είναι η πιο σύγχρονη που υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορών κρατών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα και θα πρέπει νομίζω να ανταλλάξουμε τις καλές πρακτικές. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι μια, οι διάφορες καινοτομίες στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον, ούτω ώστε να έχουμε ακόμα πιο φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές, ακόμα πιο αποτελεσματικές τεχνικές για την εξόρυξη του χρυσού. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε στην Ευρώπη για αυτά τα θέματα, ούτω ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνάδελφοι με έχουν πείσει, διότι περιέγραψαν πώς τις χώρες τις οποίες έχουν ζήσει, δηλαδή στην κομμουνιστική Τσεχοσλογαφία, υπήρχε μία ξέφρενη εκμετάλλευση και αυτή είναι που σήμερα πρέπει να προασπιστούν την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Τέτοιες ε, κινήσεις χρειαζόμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη διότι αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες. Οπότε ε, γιατί να μην ε, βρούμε κάποια λύση η οποία μας ικανοποιεί τεχνολογικά και να πούμε σαφώς ότι θα καταστρέψουμε ορισμένα πράγματα μετάκλητα και θα μας βλαστημάνε στη συνέχεια οι επόμενες γενιές. Ως εκ τούτου το αυτό που είναι βασικό είναι να έχουμε ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα και ε, να μην ε, ε, θέτουμε σε κίνδυνο τους ποταμούς οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι διασυνοριακοί. Η αλλως ειναι διασυνοριοικοί. κυρια έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να μειώσουμε τους κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από επικίνδυνες αλλά και τοξικές ουσίες ίων ή ενώσεις χιανίου. Αλλά δεν είναι πανάκια η απαγόρευση αυτών των ουσιών. Είναι επικίνδυνες αυτές οι ουσίες και χρησιμοποιούνται και σε άλλες βιομηχανικές διεργασίες και όχι μονάχα στην εξόριξη το ατύχημα της Μπάια Μάρε του 2002 δεν είναι μοναδικό. Υπήρξαν και άλλα ατύχηματα που έγιναν στην Ισπανία το 1998 και 2003 στη Σουηδία. Σουηδία. Και τα δύο αυτά ατυχήματα ήταν πολύ πιο σοβαρά από αυτά της Μπάια Μάρε. Αλλά πραγματικά ο κίνδυνος που προήλθε ήταν ο ίδιος και από τα δύο. Το 80% της παραγωγής ή παραπάνω του χρυσού γίνεται με χρήση κυανιούχων το να απαγορεύσουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει εναλλακτική τεχνολογία η οποία να είναι ε, να έχει αποδοτικότητα δεν είναι λογικό. Δεν μπορούμε να έχουμε τεχνικές οι οποίες να είναι πιο οικολογικές αλλά έχουν μεγάλο δυσβάστακτο οικονομικό κόστος. Ευχαριστώ. Κύριο Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε ο κύριος Τάκουλα προηγουμένως, οι ενώσεις Κιανίου είναι η σημερινή και αποδεκτή μέθοδος, αλλά φυσικά είναι μια μέθοδος η οποία έχει πολλούς κινδύνους. Και όπως είπε και η κυρία Μπασέσκου, ο Δούναβης έχει ήδη μολυνθεί σημαντικά από τις δραστηριότητες αυτές και εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία του να προστατεύσουμε τις ε, περιοχές οι οποίες βρίσκονται γύρω από το Δούναβη. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουμε περιορισμένη ικανότητα εξόριξης χρυσού, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει χρήση τεχνολογίας εχμής σε διάφορα μέρη. Και στη Γερμανία ακόμα έχει αναπτυχθεί μια τεχνολογία η οποία θα επιτρέψει εν καιρό να αποφύγουμε τη χρήση των ε, χιανιούχων ουσιών. Αλλά πρέπει να γίνει αποδοτικότερα αυτή η τεχνολογία, να γίνει μια τεχνολογία η οποία είναι προσιτή οικονομικά και η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε έτσι να έχουμε ένα ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την οικονομία μα. Ευχαριστώ πολύ. Μερσή, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν και ανίδιο ε, για την εξόριξη επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Διότι το κιανίδιο και οι σχετικές μέθοδοι ε, απαγορεύονται σε ορισμένα κράτη αλλά η μόλυνση των υδάτων είναι διασυνοριακή ε, και ε, το ατύχημα στην Ρουμανία επηρέασε επίσης την Τσεχοσλοβακία δεν πρόκειται για τη Ρουμανία όχι για την Τσεχοσλοβακία αλλά επηρέασε πέραν της Τσεχοσλοβακίας και την Ουγγαρία και ε, ε, ε, δημιούργησε μολύνσεις σε πέραν των χιλίων χιλιόμετρων πλήττοντας τους πολίτες που διαβίωσαν σε αυτές τις περιοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προασπίσουμε την υγεία των πολιτών και να απαγορεύσουμε τη χρήση του κιανιδίου και να υπάρξει μια ενιαία νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί του θέματος. Ο κύριος Μάτουλα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρόκειται για μια χημική ένωση που δεν είναι πολύ ελεγχόμενη και ε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν πάνω από 10.000 ε, χημικές ενώσεις και υπάρχουν ε, εκατομμύρια καταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να είναι επικίνδυνες και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Βεβαίως και το κιάνιο είναι τοξική ουσία. Είμαι χημικός ε, και μπορώ να σας πω ότι έχουμε τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Το 18% του κιανίου χρησιμοποιείται στην εξοριστική βιομηχανία, το υπόλοιπο χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία ή στην ε, βιομηχανία των καλλιντικών. Επίσης, ε, σε αυτό το πλανήτη ε, χρησιμοποιούμε ουσίες που είναι χίλιε φορές πιο τοξικές από το ωκεάνιο. Ε, βεβαίως, οι τοξικές ενώσει, όταν φτάσουν στο νερό καταστρέφουν τη ζωή. υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που καταστρέφονται από άλλε ενώσει. Παραδείγματο χάρη το ε, χλωρίχο νάτριο μερικές φορές σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι πάρα πολύ α, θανατηφόρο. Ε, και όμως το τρώμε κιόλα. Η Ρουμανία ως ευρωπαϊκό κράτος αποφάσισε λοιπόν να προβεί σε ορισμένα μέτρα να κάνει κάποιους, ε, να προβεί σε κάποιους περιορισμούς. Όλα τα κράτη θα πρέπει να ακολουθήσουν την οδό της Ρουμανίας. Κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση είναι λανθασμένη. Το θέμα που μας απασχολεί είναι πολύ περίεργο. Ε, υπενθυμίζει ένα ατύχημα που έγινε πριν από 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί αυτή η μακρά σιωπή και γιατί τώρα το θυμηθήκαμε, γιατί συζητάμε τώρα. Αν ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, τότε θα πρέπει να απαγορεύσουμε τα πάντα που συνδέονται ε, με ατυχήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητη όλη η στάση μας και χρησιμοποιούμε το περιβάλλον ως ε, ε, οθόνη καπνού. Νομίζω ότι απλώς πρόκειται για κακή ε, πολιτική, κακό πολιτικό τέχνασμα. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος πριν ζητήσω από την Επίτροπο να πάρει το λόγο, ο κύριος Πόσελτ ίσως. Πολύ σύντομα, ε, γνωρίζω πολύ καλά την Πάγια Μάρης, ξέρω ότι δεν είναι στην παλιά Τσεχοσλοβακία, αλλά βόρεια του Σιντ Μπρέτνικ υπήρξε ένα λάθος μεταφραστικό και είχα αναφερθεί στις ομιλίες της κυρίας Ρότοβας που αναφέρθηκε στην ε, εμπειρία του ο Κάπας ε, Κιχώρη. Δηλαδή γνωρίζω καλά την γεωγραφία της Κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και προφανώς θα εξασφαλίσω ότι ο κ. Ποτόσνικ θα λάβει πλήρως γνώση της συζήτησης αυτής και φυσικά συμμεζόμαστε τις ε, ανησυχίες σας για τις κιανίουχες ενώσεις. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετά από το τρομερό ατύχημα της Μπάια Μάρα η Κομισιόν έχει αντλήσει ήδη συμπεράσματα και η οδηγία που έχουμε εγκρίνει περιλαμβάνει πολλούς περιορισμούς, πολλές προϋποθέσεις, πολλές ε, αιτήσει που έχουν σε στόχο να εξασφαλίσουν ότι θα προστατευτεί το περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και η ανθρώπινη υγεία. Η οδηγία αυτή θα μειώσει και την πιθανότητα να ανακύψει και πάλι ένα τέτοιο ατύχημα και ακόμα και αν υπάρξει ατύχημα θα περιορίσει τον αντίκτυπό του προς το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η οδηγία να εφαρμοστεί πλήρως και ο πρεπόντος. Λόγω των ιδιαίτερα ε, αυστηρών προϋποθέσεων και προδιαγραφών της οδηγίας για την εξόριξη, μια πλήρης απαγόρευση της χρήσης χιανίχων ουσιών για την εξόρυξη χρυσού δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι πρόσφορη, αλλά εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές μεθόδους και θα επανέλθουμε το 2012. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλύτερη ανακύκλωση των ορυκτών που περιέχουν ε, χρυσό και των αποβλήτων για να έχουμε ανάκτηση χρυσού και να μειώσουμε την εξόρυξη. Θέλω λοιπόν να σα ευχαριστήσω. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά στον κύριο Ποτόσικ, ο οποίο νομίζω θα είναι στη διάθεσή σα να απαντήσει εν καιρό περαιτέρω ερωτήματα. Η Κομισιόνα αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με μεγάλη προσοχή, αλλά αν δείτε την οδηγία βλέπετε ότι πολλέ από τι ανησυχίε σα έχουν τύχει ήδη απόκριση και εμεί λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη πάρα πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πίτροπε ώστε αγαπητοί συνάδελφοι έχει κλείσει η συζήτηση η ψηφοφορία θα γίνει το Μάιο και πρέπει να σας πληροφορήσω ότι και αυτή η Σύνοδος Ολομέλειας έχει κλείσει. Σας εύχομαι ένα ασφαλές ταξίδι επιστροφή της χώρες σας χωρίς ηφαίστεια ή άλλες παρεμβολές. Ευχαριστώ.